Uh, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσουμε. We start votes. We start the votes. Αρχίζουν οι ψηφοφορίες, παρακαλώ. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης Αγιάλα Σέντερ με θέμα το διορισμό του κυρίου Βέσμπερκ ως μέλους του ελεκτικού συνεδρίου. Περνάμε στην ψηφοφορία του σχεδίου απόφασης. Δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες. Θα χρησιμοποιήσουμε τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας παρακαλώ και η ψηφοφορία θα είναι μυστική. Η ψηφοφορία, αγαπητοί συνάδελφοι, θα είναι μυστική. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Ο συνήθως, φυσικά. Μπορείτε να πατήσετε ναι ή όχι ή αποχή. Η μόνη διαφορά έγκυται στο ότι το μπλε φω θα φαίνεται. Δεν θα φαίνεται το πράσινο, το κόκκινο, το άσπρο, ανάλογα με το υπέρ κατά η αποχή, αλλά θα φαίνεται μόνο ένα μπλε φω γιατί η ψηφοφορία είναι μυστική. Ξεκινάμε, συνάδελφοι. Otwieram głosowanie. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ο διορισμός του κυρίου Βέσμπεργκ και συγχαίρουμε την εισηγήτριά μας, την κυρία Γιάλα Σέντερ. Περνάμε στην έκθεση Wallis, αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της κυρίας Άγνιας Χάνκης. Θα ψηφίσουμε την έκθεση. Ποιος είναι υπέρ της άρσης. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και ευχαριστούμε την κυρία Γουόλες για την έκθεσή της. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, η έκθεση Ζαχραντήλ, δικαιολογητικά καταγωγή ορισμένων κλωστιφαντουργικών προϊόντων από τρίτε χώρε. Ο κύριο ε, Ζαχράντιλ, ο εισηγητή, ήθελε το λόγο. Σα ακούμε, κύριε εισηγητά. Σύντομα μόνο, Πρόεδρε. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα όταν ορίστηκα εισηγητής. Είχαμε την ευκαιρία ε, να καταργήσουμε ένα νομοθέτημα και να μην το δεχτούμε. Ε, είναι ε, περίτο και αυτό που έχουμε ως μακροπρόθεσμο και πάγιο στόχο είναι το εφνομοθετήν. Ε, οπότε ε, σας παρακαλώ να υποστηρίξετε την κατάργηση αυτής της νομοθεσίας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Σας ευχαριστώ. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση την έκθεση του κυρίου Ζαχραντήλ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Ζαχαραντήλ. Περνάμε στην έκθεση Σερακιάνη για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας σε εργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Η κυρία Ντεκάιζερ ζήτησε το λόγο. Ξέχασα την κάρτα μου. Έτσι. Uh, Εντάξει συνάδελφοι. Ε, πω. Τεράστιο πρόβλημα για όλους μας. Έκθεση τη κυρία Σερακιάνη για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας σε εργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Σερακιάνη. Έκθεση Οκονή για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης ευρώ. Η κυρία εισηγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ως εισηγήτρια και εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων που συμφωνούν, ζητώ αναβολή της ψηφοφορίας των δύο εκθέσεων που αφορούν της μεταφοράς ευρών σε μετρητά. Είναι η παρούσα έκθεση και μια άλλη λίγο πιο κάτω, η έκθεση της Επιτροπής ε, Εξωτερικών 076. Ε, ε, Είναι για λόγους διαδικαστικούς για καλύτερη συνεργασία Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συμβουλίου. Παρακαλώ να ψηφίσετε αναβολή της έκθεσής μου και της επόμενης έκθεσης πάλι δικής μου. Σας ευχαριστώ. Έχουμε δύο αιτήματα. Θέλουμε κάποιον που να υποστηρίξει αυτή την πρόταση. Θα ακούσουμε δύο ε, παρεμβάσεις υπέρ και κατά κύρια Μπόλης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής. Ε, ζήτησε η Επιτροπή μας να αναβληθεί αυτό, οικονομική, γιατί ε, έχουμε ένα πρόβλημα στη διαδικασία. Στο κείμενο του κειμένου, μια αιτιολογική σκέψη που είχε συμφωνηθεί σε μια γραπτή διαδικασία ε, ε, τριμερούς, διαλόγου αφαιρέθηκε και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς γιατί ήταν γραπτό. Μας είπαν ότι διαφωνεί η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου ε, γιατί ε, δεν συνάδει πλήρω με την κοινή ε, συνεννόηση. Η κοινή συνεννόηση δεν είναι νομική βάση και σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε κάτι τέτοιο ω προηγούμενο και δεν θα ψηφίσουμε μέχρι να λυθεί το ζήτημα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η διοργανική συμφωνία ή η κοινή συνεννόηση ή οτιδήποτε άλλο να περιορίζει τις εξουσίες του Κοινοβουλίου που απορρέουν από τη συνθήκη. Οπότε δεν μπορούμε ε, να το δεχτούμε. Αυτό θα αποτελέσει προηγούμενο και θέλουμε να ε, ξεκαθαρίσουμε προς όλες τις ότι δεν είμαστε πρόθυμοι να το δεχτούμε. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς να μιλήσει εις βάρος του αιτήματος της ηγετρίας της κυρίας Οκονή. Όχι. Άμα. Ο κύριος Περώνη. Πρόεδρε ουσιαστικά δεν είμαι κατά της πρότασης, αλλά τη Δευτέρα το απόγευμα επίκειται η έγκριση, μάλλον εγκρίνουμε ε, την διάταξη των εργασιών για όλη την εβδομάδα και διερωτώμε γιατί δεν έγινε αυτή η πρόταση αναβολής εχθές και γίνεται ε, σήμερα πάνω στη ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε την πρόταση της κυρίας Οκονή. Ποιο είναι υπέρ της προτάσεως Σοκονή για αναβολή. Κατά αποχές εγκρίνεται, οπότε αναβάλλονται και οι δύο ψηφοφορίε ε, των εκθέσεων της κυρίας Σοκονή. Επόμενη έκθεση, έκθεση Τσίκαου για τι εφαρμογέ του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης Μεταφορές. Ψηφίζουμε ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Τσίκαου. Έκθεση Σίμψον. Διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Σίμψον. Έκθεση Ελχαντράουι. Δεύτερη ανάγνωση. σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σε ό,τι αφορά την επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα. Έκθεση ε, πρόταση του Συμβουλίου θα πρέπει να συγκεντρώσουμε ενισχυμένη πλειοψηφία. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματο. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Συμφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οπότε η ούτως σε θέση του Συμβουλίου έγινε δεκτή. Και συγχαίρω τον κύριο Αλχαντράουι, τον εισηγητή. Έκθεση Λάινεν τώρα. Ευρωπαϊκή περιβαλλοντοοικονομική λογαριασμή έκθεση του σχεδίου κανονισμού. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροποποιήθηκε λοιπόν η πρώτη της Επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται και η τροποποίηση του κειμένου της Επιτροπής. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, χωρίς τροπολογίες. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Λάινεν. Περνάμε στη δεύτερη έκθεση Οκονή που έχει αναβληθεί και αυτή, μην το ξεχνάτε. Οπότε περνάμε στην έκθεση Οντί για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης. Έκθεση ψηφίσματος χωρίς τροπολογίες. Ψηφίζουμε το 21. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 18 και πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 24 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 47. Σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ. Ο κύριος Κόβαου. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ενημερώσω τη γραμματεία ότι έχω προφορική τροπολογία για τη διαγραφή του άρθρου 27 γιατί το άρθρο αυτό περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες σε ό,τι αφορά σημαντικό, το σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα INDECT. Θα ήθελα να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι το πρόγραμμα αυτό έχει την έγκριση του Ethical Review. Έγινε στις 5 Μαρτίου του 2011 η εξέταση από εμπειρογνώμονες της Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας και ε, έχει εγκριθεί το σχέδιο, ήταν θετική η εξέταση. Δεν, δεν υποβλήθηκαν επιφυλάξεις. Οι ιδεοντολογικές πτυχές του σχεδίου αυτού τυχάνουν του συνεχούς ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από την αρχή. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω το Κοινοβούλιο να εξετάσει αυτό το ζήτημα και να παρακαλέσω να διαγραφεί το σχετικό άρθρο. Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουμε στην έκθεσή μας ανακριβείς πληροφορίες και αβάσιμες επιστημονικά είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η επιστημονική κοινότητα από όλη την Ευρώπη και έδρα ε, βρίσκεται στην Κρακοβία. Έχει υποβληθεί προφορική τροπολογία κυρίες και κύριοι που ζητά την διαγραφή ολόκληρης παραγράφου 27. Ερώτηση πρώτη. Έχει κανείς αντίρρηση. Θα παρακαλούσα να σηκωθούν όσοι έχουν αντίρρηση. 40 ευρωβουλευτές, άρα δεν πρόκειται να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία, η οποία καταπίπτει. Επαναλαμβάνουμε 47 παράγραφος σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος? Κατά αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 60. Ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σχέση ε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. E, e, Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ πρέπει να εκενώσετε την αίθουσα, σπεύστε προς την κοντινότερη θύρα. Πρέπει να σπεύσετε στην κοντινότερη σας έξοδο. Μην χρησιμοποιήσετε τα ασανσέρ και μην επιστρέψετε στα γραφεία σας παρακαλώ. Μην επιστρέψετε στα γραφεία σας. Και εγκαταλείψτε το κτίριο το συντομότερο δυνατόν. Επαναλαμβάνω, εγκαταλείψτε το κτίριο το συντομότερο δυνατόν. Και μην επιστρέψετε στα γραφεία σας. All of us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 Ε, θα ήλπιζα ότι θα ήξερα τι γίνεται με τις επεξηγήσεις ψήφου. Ευχαριστώ πολύ.